zetten. Veo que podemos decir colegas, porque hasta hace un momento solo había uno, pero ahora ya podemos hablar en plural. Θέλουμε να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας αυτή τη στιγμή. Η μερισσία διάταξη προβλέπει να εξετάσουμε την έκθεση του κύριου Σίβη πάνω στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα.